Ε, η σοσιαλιστική ε, ομάδα μου έστειλε αίτημα για τον ορισμό του κυρίου Νταλή στην Επιτροπή Αναφορών. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επιβεβαιώνεται αυτός ο ορισμός. Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη.